Χρειάζεται διάλογος, είπατε, στην ομάδα Βίσεγκραντ. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω όμως κατά τη γνώμη σας ποιο είναι το καθοριστικό χαρακτηριστικό της Κεντρικής Ευρώπης και πώς πρέπει εκείνη να συνομιλεί με την υπόλοιπη Ευρώπη. Λόπες Αγγελάρ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρωθυπουργέ Μπελεγκρίνη, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και που μιλήσατε για περισσότερο κοινωνική Ευρώπη, για ίσους μισθούς, ε, καταπολέμηση της ανεργίας. Ε, ωραία, ό,τι καλύτερο να τα καταφέρετε. Και για τον υποψήφιο για τη Σλοβακική Προεδρία. Ελπίζω επίσης να καταφέρετε να διερευνήσετε την δολοφονία των δημοσιογράφων και να καταπολεμήσετε τη διαφθορά σε βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Για την ομάδα του Βίσεγκρου, ποια είναι η φύση του, για ποιο λόγο υπάρχει. Και το πιο σημαντικό, το ακούσατε από πολλούς από εμά που λένε ότι στόχος της ομάδας Βίσεγκρουπ είναι να κλείσουν τα εξωτερικά σύνορα προκειμένου να αποφύγουμε τον εξισλαμισμό και τη σαριά. Εσείς συμφωνείτε με αυτήν την βλασφημία ή διαφωνείτε με αυτό, γιατί δεν το ακούσαμε, δεν αντιδράσατε όταν ακούσατε τέτοιες προσβολές. Είναι Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας Βίσεγκριτ. Βίσεγκρατ, παρακαλώ να μας απαντήσετε κύριε Πελεγκρίνη. Ο κύριος Σαρμπάτη τώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτά που είπατε αποτελούν και μια απάντηση στα όσα ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Όπως και εσείς, είπε και εκείνος ότι χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ε, ευρωπαϊκά καθορισμένο κατώτατο μισθό. Γνωρίζουμε όλοι ότι το επίπεδο τη ευημερία είναι εκείνο που καθορίζει το επίπεδο των επιδομάτων. Επειδή όμως εντός Ευρωπαϊκή Ένωση το επίπεδο της ευημερίας είναι ε, διαφορετικό. Δεν, μπορούν να υπάρξει, δεν μπορεί να υπάρξει ενιαίος κατώτατος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό θα δημιουργήσει ανεργία. Υπάρχει άνηση κατανομή του πλούτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θέλω να παραθέσω από αυτό που είπε ο Μακρόν. δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστική κρίση αν δεν είχαμε το ευρώ. Δεν υπάρχει πιο λανθασμένη δήλωση από αυτήν, διότι το ευρώ δεν ενίσχυσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, την αποδυνάμωσε και τη δίχασε. Το, ε, η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή παρουσιάζει σε ολόκληρο τον κόσμο το χαμηλότερο ποσοστό ανάπτυξης και μεγένθησης. Είναι fake news αυτά. ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, Πρωθυπουργέ. Η παρέμβασή μου θα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος. Σκεφτόμουν ότι θα μας πείτε ποιο είναι το πραγματικό σας όραμα. Ότι θα έρθετε σαν Πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Πρωθυπουργός μιας κυρίαρχη χώρας, να μας πείτε για τη μεταρρύθμιση, να μεταρρυθμίσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως παραδείγματος χάρη την κοινή αγροτική πολιτική. Ξέρετε ότι μπορείτε να καθορίσετε το πού διατίθενται οι πόροι γεωργικοί. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα θέλω να θέσω και θα ήθελα απάντηση. Οι συνάδελφοι εδώ ανέφεραν θύματα βιοπραγιών στη Σλοβακία. Βλάντο Ρίμπαρ. Ο Βλάντο Ρίμπαρ ήταν γεωργό. Το συναντήσαμε όταν πήγαμε στην Πρατισλάβα. Είχε ένα αγρόκτημα, όχι πολύ μακριά, και μα είπε στην ομέτα φτάσαμε ότι είχε αυτοκτονήσει. Τώρα φαίνεται ότι δολοφονήθηκε ο Βλαντό Ριμπάρ. Ερώτηση εξηχνιάζεται και, αυτού, και αυτή η υπόθεση. Εξεχνιάζονται και τέτοιου είδου υποθέσει. Θα βρεθεί η λύση, η απάντηση. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτή την υπόθεση και θα ενημερώσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θέλει να απαντήσει αμέσω ο Πρωθυπουργό ο κ. Πελεγκρίνη. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω αμέσως, γιατί δεν θα ανεχτώ τέτοιου είδους ε, συκοφάντηση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σηκώνεται δηλαδή ένα μέσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκτοξεύει τέτοιου είδους ψεύδι. Αναφερθήκατε στον κύριο Ριμπάρ και θέλετε να δημιουργήσετε την εντύπωση ότι δολοφονήθηκε λόγω ε, ζητημάτων που, που σχετίζονταν με τα αγροτικά κονδύλια και τις επιδοτήσεις. Να σας πω τι είπε ο ίδιος ο γιος του. Ο γιο του είπε ότι τον εκμεταλλεύτηκαν τον κύριο Ριμπάρ άνθρωποι που δεν του είχε συναντήσει ποτέ και που εκμεταλλεύονται την μνήμη του διοργανώνοντας διαδηλώσει. και ότι δεν θα ήθελε κανένα να εκμεταλλεύεται τον θάνατο του πατέρα του. Δεν θέλει κανείς να καταχράτε τη μνήμη του πατέρα του για πολιτικό όφελος. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω να σταματήσετε να δεσπείρετε φήμες ψευδείς για τη Σλοβακία. Έχετε κι εσείς προβλήματα στην ε, Τσεχία, εγώ όμως ποτέ δεν έχω πει τέτοιου είδους ψέματα για τη χώρα σας. Αν θέλετε δηλαδή να έχουμε μια ίση και ισότιμη ε, συζήτηση. Ε, αγροτικές επιδοτήσεις και ταμεία. Εγώ έχω μιλήσει για αυτό το θέμα και έχω δηλώσει ότι χρειάζεται πράγματι να αλλάξουν οι κανόνε και να μην χρηματοδοτούνται οι άνθρωποι που απλώ στα χαρτιά έχουν γεωργικέ εκτάσει τι οποίε δεν δουλεύουν. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα ταμεία αυτά θα πηγαίνουν σε ανθρώπου που πραγματικά εργάζονται και δουλεύουν τη γη και όχι το αντίθετο. Nord Stream. Ναι. Ακούστηκαν πολλά όμορφα λόγια για το πώς πρέπει και μπορούμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Ναι, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε μια υπόθεση όπου μπορούμε άθελά μας να βλάψουμε ε, ανθρώπους. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να παράσχουμε φυσικό αέριο στην ε, Ουκρανία φέτος το χειμώνα για να εξασφαλίσουμε και να συμβάλλουμε στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αυτής. Όμως η ιδέα ότι θα πρέπει να ε, φροντίσουμε την Ουκρανία είναι κάτι το οποίο βεβαίως βρίσκει ευήκο αότα και στους, ε, επιχει... στους, επιχειρήσεις... στους επιχειρηματίες της Ουκρανίας. Όσον αφορά την, ε, την έδρα του της... και την κατανομή της ε, αρχής εργασίας, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, δύο συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε αυτό. Ε... Είπαν κάποιοι ότι οι νέοι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν την έδρα του στα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα ε, οργανισμούς. Τελικά όμως ε, οι οργανισμοί αυτοί ε, κατέληξαν σε παλιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη-μέλη τα οποία ήδη φιλοξενούσαν ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Όταν λοιπόν μιλάμε για την υπέρβαση της, του διαχωρισμού ανάμεσα στην Ανατολή και τις Δύσεις, να ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Εγώ πάντοτε με ανοιχτό πνεύμα απαντώ ε, στα ερωτήματά σας. Συνάθε Τόμασιτς. Ευχαριστώ τον ε, Πρωθυπουργό Μπελεγκρίνη. σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να συνεισφέρετε στη συζήτηση αυτή για το μέλλον τη Ευρώπη. Σίγουρα η Σλοβακία θα έχει καλά αποτελέσματα. όπω είπατε και εσεί, τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα. Ο δρόμο μερικέ φορέ ήταν δύσκολο, αλλά η Σλοβακία είναι πιο προχωρημένη από ό,τι ήταν ε, όταν απέκτησε την ανεξαρτησία τη. Έχει πάρει το μέλλον της στα χέρια της και αυτό βοηθάει στην ευημερία του λαού της, καλύτερη ποιότητα ζωή εκεί. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι η ανεξαρτησία ήταν το σωστό για τη χώρα σας. Όμως τώρα συστήνεται μια μεγαλύτερη πολιτική ολοκλήρωση. Δηλαδή λέτε ότι οι αποφάσεις για τη Σλοβακία, το μέλλον της Σλοβακίας πρέπει να πάει σε χέρια πιο συνολικά και με κοινέ αξίες, ε, με αδελφότητα κτλ. Άρα τελικά μπαίνουμε σε μια διαφορετική λήψη αποφάσεων, διαφορετική διαδικασία, όπου μικρότερες χώρες όπως η δικιά σας η χώρα, η δικιά μου, μπορούν λιγότερο να προστατεύουν τα δικά του συμφέροντα. Μα η συγκέντρωση τη εξουσία της Βρυξέλλε δεν μπορεί να συμφέρει ούτε το ούτε την Πρατισλάβα. Ευχαριστώ. Σούρικ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Η Σλοβακία έχει σίγουρα πολλά δικά της προβλήματα, τη μαφία, τη διαφθορά και τα περισσότερα από τα προβλήματα αυτά πρέπει να λυθούν σε εθνικό επίπεδο. Από μια κυβέρνηση η οποία να είναι εκλεγμένη με ανοιχτές, ελεύθερες εκλογές και μυστική ψηφοφορία. Θα ήθελα να υποστηρίξω ε, να σας υποστηρίξω κατά της, ε, των κατηγοριών που ακούστηκαν. Ε, είναι άδικο ο κύριος Παπαδημούλης να δίνει μαθήματα στη Σλοβακία όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική. Υπάρχει η διερεύνηση για τη δολοφονία των δημοσιογράφων. Αυτό γίνεται, ακούστηκε. Και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Κρέσλερ για τις δικές της προσπάθειες. Τώρα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να μειώσει το διχασμό ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, μια στιγμή να βάζουμε τα ίδια κριτήρια για όλους, να πληρώνουμε τις ίδιες επιδοτήσεις σε όλους, να δούμε ποιος ε, τελικά παραβιάζει τις κυρώσεις για τον Nord Stream 2. Τότε θα υπάρχει ισότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας υπέρ της κοινωνικής Ευρώπης και για την προσπάθεια που κάνετε υπέρ του ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού. Αυτό που τόνισε μόλις και ο πρόεδρος Γιούγκερ. Οι πολιτικές ε, που εφαρμόστηκαν στη Γερμανία από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ε, πραγματικά ωφέλησαν ιδίως τους ανθρώπους στην Ανατολική Γερμανία. Όμως ε, βλέπετε ότι οι συντηρητικοί κρατούν αποστάσεις. Η νέα πρόεδρος των χριστιανοδημοκρατών στην Γερμανία μίλησε αρνητικά ε, και διαφώνησε με την πρόταση ε, θέσπισης κατώτατου μισθού. Ξέρετε όμως ότι έχει πάρα πολύ σημαντικά. Αυτή τη στιγμή εσείς ηγείστε της ομάδας του Βίσεγκραντ. Σας ως Ανατολικό Γερμανός, ως Γερμανός του Βίσεγκραντ, σας καλώ να το ξεκαθαρίσετε αυτό και στην ε, Ουγγαρία και στην Πολωνία. Μαζί καταπολεμήσαμε το σοσιαλισμό. Παρακαλώ να κάνουμε όλοι μαζί από κοινού προσπάθειες για την Ευρώπη που θέλουμε. Σκρίπεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μα παρουσιάσατε το όραμα για την Ευρώπη, για τη Σλοβακία και για τη Σλοβακία στην Ευρώπη. Συμφωνώ μαζί σα, ότι η Σλοβακία θέλει να είναι ένα υπεύθυνο εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ελοκλήρωση και στην λειτουργία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Θέλουμε όμω πραγματικά να είμαστε μέρο όλων των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι θέλετε να βρίσκεστε στην καρδιά των εξέλιξεων. Θέλετε όμως περισσότερη Ευρώπη όσον αφορά τον κοινωνικό πυλώνα ή τον Ευρωστρατό για παράδειγμα. Εγώ ως Σλοβάκος Ευρωβουλευτής πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε για την ανάγκη να μειωθούν οι παρεμβάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς που εμπίπτουν στο, στην επικουρικότητα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν περισσότερες προσπάθειες εκεί όπου πραγματικά οι ευρωπαϊκές, οι κοινές ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκές αξίες μπορούν να ενισχυθούν. Πρέπει να ενισχύσουμε τις ευρωχριστιανικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε η Σλοβακία να αποτελεί ένα ισχυρό τμήμα και εταίρο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να συνεργαστούμε ε, με όλους ώστε να εξασφαλίσουμε το μέλλον της Ευρώπης. Ολοκληρώθηκε το ΚΑΤΣΔΙΑ. Δίνουμε το λόγο στον Πρωθυπουργό τη Δημοκρατία τη Σλοβακίας, τον κύριο Πελεγκρίνη, για να απαντήσει στις τελευταίες ερωτήσεις που του ετέθησαν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Προτού περάσω στις ε, καταληκτικές μου παρατηρήσεις, θα ήθελα να απαντήσω σε μια ερώτηση που μου απευθύνθηκε εδώ. Ποιος είναι ο ρόλος και ποιος είναι ο χαρακτήρας, ποιος είναι το καθήκον της Σλοβακίας και της ομάδας των χωρών του Βίσεγκραντ εγώ θα το επέκτηνα το ερώτημα. Ποιο είναι το καθήκον όλων των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθήκον είναι ένα και μοναδικό. Να εξασφαλίσουμε την ευημερία των ε, πολιτών των χωρών μας. Αυτό είναι ο βασικός και κύριος στόχος βάσει του οποίου αναλαμβάνουμε τα καθήκοντά μας. Η ευημερία των πολιτών. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας κάνω έκκληση. Να υπάρχει σεβασμός. Ή θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί. Έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός της ευημερίας όλων των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκεί και πέρα μπορούμε να περάσουμε και σε ε, άλλα θέματα. Πώς μπορείτε να αναφέρεστε σε ψευδοζητήματα όπως αυτά που αφορούν ε, ε, τους ε, ηλικιωμένους. Θεωρώ ότι δεν έχουμε κάνει όλα όσα έπρεπε για να, επιτευχθεί αυτός ο στόχος της ευημερία όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι έχουμε βελτιώσει τους όρους διαβίωσης των πολιτών μας στις περιοχές των ε, χωρών μας Πραγματικά είμαι περήφανος για τα όσα έχουμε καταφέρει και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές που ε, υπερασπίστηκαν και υποστήριξαν την ε, δημοκρατία της Σλοβακίας μέσω των τοποθετήσεων τους. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι να πω τα εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει για τη Σλοβακία και για τον πυλώνα της ελευθερίας και της ε, ε, ε, ευημερίας πολύ σημαντικός εταίρος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, ελλείψεις, γνωρίζουμε ότι αντίστοιχες ελλείψεις και ελλείμματα υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε όμως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο να υπερβούμε τα προβλήματα. Θέλουμε να συνεργαστούμε για κοινωνική πρόοδο, για προστασία του περιβάλλοντος, για οικονομική ανάπτυξη και εδώ πραγματικά ε, πρέπει να επιδιώξουμε την ενότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντική η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω. Μιλήσαμε για την ε, πολιτική συνοχής. Η πολιτική συνοχής θεσπίστηκε ώστε να μπορέσουμε να υπερβούμε μεγάλες περιφερειακές ανισότητες όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και εντός του κάθε κράτους μέλους. Εδώ η πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να γίνει όμοιρος της ε, ευρύτερης, της γενικής πολιτικής. Το να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή την, τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής νομίζω ότι δεν είναι σωστή η ιδέα. Η πολιτική συνοχής υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει ακριβώς διότι υπάρχουν περιφερειακές ανισότητες και στόχος και καθήκον μας είναι να ξεπεράσουμε τις ανισότητες αυτές. Αν επιτευχθεί ο στόχος αυτός μπορούμε να ξανασυζητήσουμε το αν χρειαζόμαστε την ε, πολιτική συνοχής. Επαναλαμβάνω λοιπόν την έκκλησή μου. Στόχος μας είναι να φέρουμε όσο πιο κοντά ε, σε εμάς, στους, ε, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τους Ευρωπαίους πολίτες. Εγώ από την πλευρά μου δεσμεύομαι ότι θα κάνω ό,τι περνά από, τα, από το χέρι μου ώστε η Σλοβακία να παραμείνει μια θετική επικοδομητική δύναμη της κεντρικής Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου τιμή που βρέθηκα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Κύριε Πρωθυπουργέ, διακόπτουμε για λίγα λεπτά και μετά θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε σε λίγο την ψηφοφορία σε 30 δευτερόλεπτα, οπότε παρακαλώ ετοιμάστε τις κάρτες σας. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε την ψηφοφορία τώρα. Καθίστε παρακαλώ. Πρώτη έκθεση. Υπάρχει ένα διαδικαστικό όμως, αλλά για να δω. Η κυρία Πιλτσέρνου, παρακαλώ. Θα ήθελα πριν περάσω στην ψηφοφορία να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου την αδικία ε, που, που ε, το βραβείο Ζαχάροφ καταδικάστηκε, καταδικάστηκε σε τέσσερις δεκαετίες φυλάκιση σε 148 μαστιγώσεις διότι υπερασπίστηκε στο Ιράν τα δικαιώματα των γυναικών που ζήτησε στο Ιράν την κατάργηση της θανατικής ποινής. Πιστεύω ότι αυτό το κοινοβούλιο, Πρόεδρε, μέσω της φωνής σας και του Προέδρου του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να εκφράσει άμεσα μια καταδίκη, απόλυτη καταδίκη έναντι αυτής της επονίδης της καταδίκης που σημειώθηκε στο Ιράν και θα πρέπει να ζητήσουμε αμέσως να απελευθερωθεί άμεσα ανεφόρον η Ναστρίν Σοτουντέ. Διότι είναι απίστευτο το Ιράν να δείχνει ακόμα μια φορά ότι είναι εχθρός, ακραίος εχθρός των δικαιωμάτων των γυναικών. Ε, και αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να τον εχθούμε, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Σημειώνουμε τα σχόλιά σας και θα τα μεταφέρουμε στον Πρόεδρο. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Έτηση του κύριου Καβαντά. Έτηση άρσης της ασυλίας της Μόνικα Χολμάιερ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Επόμενη έκθεση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 Αν ε, με το άλοθη κάποια ιδεολογία ψηφίσετε για τη φορά κατά τη Ασυλία του Ζαμαρί Λεπέν, σημαίνει ότι βρίσκεται φυσιολογικό να ελέγχετε η δουλειά των βοηθών σας, διακόπτη πρόεδρος, ο διακόπτη πρόεδρος στην ομιλήτρια. Περνούμε στην ψηφοφορία. Δεν συζητούμε τώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ψηφίζουμε την αίτηση άρσης ασυλίας του Ζαν Λεπέν τώρα. Μια στιγμή. Ακούστε με, συνάδελφοι. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Ο κύριο Καβαντά, παρακαλώ. Κύριε Καβαντά, έχετε το λόγο. Πολύ σύντομο θα είμαι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ε, μιλάμε για κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ακριβείς και να μην ε, μιλάμε κατά προσέγγιση. Η κυρία Χολμάγερ η ίδια ζήτησε την άρση της κοινοβουλευτικής της ασυλίας για ε, ένα οδικό ατύχημα. Οπότε δεν δέχομαι να μπερδεύουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση, λέει Ψηφίζουμε τώρα την ε, αίτηση άρσης Ασελίας του Ζαν Μαρί Λεπέν, έκθεση Κώστα Χρυσόγων. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τώρα πάλι αίτηση άρσης Ασελίας, Ντομινίκ Μπίλντε. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πριν περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία, η κυρία Τόμασιτς θέλει να πει κάτι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Στο σώμα αυτό ακούμε διάφορα σχέδια για την Ευρώπη, περισσότερη πολιτική παρέμβαση, περισσότερους κοινού θεσμούς, περισσότερα χρήματα για φιλόδοξα προγράμματα, Ηνωμένε Πολιτείες Ευρώπης κλπ. Μεγάλες ιδέες, αλλά τελικά πού καταλήγουν όλα αυτά. Στην επόμενη θητεία θα υπάρχουν ε, Κροάτες ε, βουλευτές. Παρόλα αυτά τα κροατικά δεν θα χρησιμοποιούνται πλήρως στις εργασίες του σώματος αυτού. Το άρθρο 159 του κανονισμού πράγματι επιτρέπει αναβολή της πλήρης κάλυψης των Ιρλανδικών, των Κροατικών κλπ και την επόμενη θητεία δεν θα μπορούμε να έχουμε ούτε πλήρη διερμηνία ούτε πλήρη μετάφραση. Μα πόσοι αιώνε χρειάζονται για να διασφαλιστεί αυτή η υπηρεσία πλήρω τα, η Μάλτα, η Ιρλανδία δεν έχουν μόνο μία επίσημη γλώσσα. Τα κρατικά Όμω, έχουν μία μόνο επίσημη γλώσσα. Οπότε πώ θα γίνει αυτό ο περιορισμό. Αγαπητοί συνάδελφοι, α προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο είμαστε όντω ενωμένοι μέσα στην ποικιλομορφία σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σα. Νομίζω ότι... Έχουμε συζητήσει αρκετά για αυτό το θέμα. Τώρα θα ψηφίσουμε για την επέκταση του άρθρου 159 του κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ε, ένα της κοινοβουλευτικής περίοδου υπέρ, κατά, αποχές. Θέλω να το ελέγξω ηλεκτρονικά παρακαλώ, οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε, πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ. Περνάμε στην έκθεση Σμιτ. Κυρία Σμιτ, όχι. Εσείς έχετε διαδικαστικό. Μια στιγμή. Κύριε Κόμπερν, θα σας δώσω το λόγο σε λίγο. Παρακαλώ, ακούστε. Παρακαλώ, κύριε Κόμπερν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν ελέγχεται με δορυφόρους, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό στα σύνορα με τη Βόρεια Ιρλανδία. Μπορεί να γίνει με δορυφόρους. Αφού το κάνουμε αυτό, σε ένα άλλο σωρό σημείο του κόσμου, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να χρησιμοποιήσουμε δορυφόρου στα σύνορα με τη Βόρεια Ιρλανδία. Πρόεδρο, κύριε Κόμπερν, δεν ε, έχω χρόνο να σα απαντήσω γιατί πάνω σε αυτό που ρωτήσατε, γιατί έχουμε ψηφοφορία. Είμαστε μέσω ψηφοφορία. Αλλά σα άκουσα. Εκτό μικροφώνου παρέμβαση του κύριου Κόμπερν. Αγαπητοί συνάδελφοι, αφήστε το συνάδελφο να μιλήσει. Τώρα τελείωσε. Συνεχίζουμε έκθεση τη κυρία Σμιτ για ηλεκτρονικέ πληροφορίε σχετικά με τι εμπορευματικέ μεταφορέ. Η νέα ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλο τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τελείωσε η πρώτη ανάγνωση λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Περνάμε τώρα στην έκθεση Χαουτάλα. Ε, θελοντική Συμφωνία Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή τη δασική νομοθεσία. Ε, ηλεκτρονικά ψηφίσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλο τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Δεύτερη έκθεση της κυρίας Χαουτάλα, πάλι ε, θελοντική συμφωνία για την, ε, το ψήφισμα, ηλεκτρονικά πάλι, ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε το πρωτόκολλο και την τροποποίηση τη Σύμβαση για την Προστασία των Ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα έκθεση του κυρίου Νόγκε η ηλεκτρονικά ψηφί ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Έκθεση τη κυρία Κάφμαν, εξουσιοδότη στα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικού αγώνε και άλλε αθλητικέ διοργανώσει. Ονομαστική ψηφοφορία μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλο τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Επόμενη έκθεση του κύριου Ασή. Πρωτόκολλο τροποποίηση συμφωνία με την Κίνα για τι θαλάσσιε μεταφορέ. Προσχώρηση τη Κροατία. Ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλο τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Έκθεση τη κυρία Μανέσκου, Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεση με την Αίγυπτο μετά την προσχώρηση Κροατία. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλο τη ψηφοφορία. εγκρίθηκε. Δεύτερη έκθεση της κυρίας Μανέσκου, Συμφωνία Εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκμενιστάν. Προσωρινή έκθεση, μονομαστική ψηφοφορία, ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην έκθεση Σκρίπεκ, εκτελεστική απόφαση για την έναρξη τη αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε, παρακαλώ. Τέλο τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Έκθεση του κ. Ντάλταν. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επικόστριτων τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου. Εκκρίς. Προσωρινή συμφωνία, 35 τροπολογία. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Το Κοινοβούλιο λοιπόν ολοκλήρωσε έτσι την πρώτη του ανάγνωση. Δεύτερη έκθεση Ντάλτον. Α, συγγνώμη, κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Έχει ένα διαδικαστικό. Παρακαλώ. ψηφίζουμε το πρώτο κομμάτι ενός συνόλου εκθέσεων που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των Ευρωπαίων και θα συμπεριλάβουμε εδώ και την έκθεση για την ουσία της εσωτερικής ασφάλειας. Είναι μια ευκαιρία να επενθυμίσουμε ότι χτες συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από τη σφαγή με τεράστιο αριθμό θυμάτων στην Ισπανία. Ήταν 11 Μαρτίου του 2004. Είναι μια καλή ευκαιρία ψηφίζοντας να περάσουμε αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης για τα θύματα της τρομοκρατίας και να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Στηρίζουμε αυτό που είπατε. Περνάμε λοιπόν τώρα στο κεντρικό σύστημα τοπισμού των κρατών μελών. Παρακαλώ. Θέλετε το λόγο. Με προλάβατε. Εντάξει, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω, βάσει του άρθρου 59, παράγραφος Γ του κανονισμού, πρώτα να ψηφίσουμε τις τροπολογίες και θέλω επίσης να ζητήσω ονομαστική ψηφοφορία για αυτή την απόφαση διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντάλτον τώρα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, διαπραγματευτήκαμε τέσσερα χρόνια. Έχουμε μια συμφωνία. Έχει κάνει υποχωρήσει στο Κοινοβούλιο. Αν περάσει κάποια τροπολογία, τότε καταπίπτει η απόφαση. Γι' αυτό είμαι κατά τη πρόταση τη Γκουε και προτείνω να ψηφίσουμε απευθεία τη συμφωνία. Πρόεδρο, ωραία. Τότε θα ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία το αίτημα του κύριου Ντεγιόγκ. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Συνεπώς, ψηφίσουμε την τροπολογία 104 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλο της ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Επόμενη έκθεση. Σροϊντοβα. Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Εδώ έχουμε διάφορες τροπολογίες. Υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 197 τώρα, με ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 172 τώρα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 199. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 174D και 191D. Με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 200 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 57, συγγνώμη διορθώνει πρόεδρος, 59 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 175D υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 177 d υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά, 179 επαναλαμβάνει πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 180 d υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 181 d υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 87 και 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 210 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 211 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 212 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 202 ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 213 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 203 ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 185 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 165 καταπίπτει. 193 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 167 δι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 195 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 169 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 207 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 171, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Ψηφίσουμε τώρα την πρόταση επιτροπής με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Και εγκρίθηκε. Το Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε έτσι την πρώτη του ανάγνωση. Επόμενη έκθεση τη κυρία Νίμπλερ όσον αφορά την πράξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλεια στην κυβερνοχώρο. Τροπολογία 258, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Το Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση. Πάμε στην έκθεση του κ. Δεκάστρο. Αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ στι σχέσει μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Τροπολογία 142, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, με την έγκριση του 142 ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρώτη ανάγνωση και δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ντεκάστρο. Εδώ είμαι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πραγματικά όλου του συναδέλφου για την εξαιρετική συνεργασία που οδήγησε στην έγκριση με τόσο ευρύ επιστήριξη τη οδηγία. Χωρί αυτό το θεμελιώδε ομαδικό παιχνίδι, δεν θα καταφέραμε σήμερα να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που μπορούσε να φανεί δύσκολο, αν όχι ανεπίτευκτο. Οι συνάδελφοι πέρασαν μόνο 11 μήνε από την παρουσίαση τη προτάσεω και σήμερα μπορούμε επιτέλου να πούμε ότι δώσαμε μια απάντηση συγκεκριμένη στα αιτήματα των γεωργών, των παραγωγών των καταναλωτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που επί μακρό χρόνων παρέμειναν χωρί να έχουν εισακουστεί. Αυτό το Κοινοβούλιο, Πρόεδρε, έκανε ένα μικρό θαύμα. Αλλά είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. Τώρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα που επιτεύχθησαν να εγγυηθούμε μια δίκαιη εφαρμογή στα κράτη-μέλη μα. Αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε, μια Ευρώπη η οποία υποστηρίζει τι πιο αδύναμε επιχειρήσει και προστατεύει του καταναλωτέ μα με προδιαγραφέ διαφανή που εξασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων και την βιωσιμότητα των παραγωγικών διαδικασιών. Πραγματικά εύχομαι ότι αυτή ε, η κατεύθυνση ακολουθεί και στο μέλλον με την ίδια προσπάθεια, με την ίδια σοβαρότητα και συνεργασία από την πλευρά όλων. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ. Πάμε στην έκθεση του κυρίου Σόπφλιν όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η κυρία Σπινέλη έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα ήθελα να παρουσιάσω εν ονόματι της ομάδας μου ένα αίτημα να ψηφίσουμε τις τροπολογίες σύμφωνα με το άρθρο 59 του εσωτερικού κανονισμού και ζητώ η ψήφος να λάβει χώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Πιστεύω ότι το παρόν κείμενο έχει κάποια λατώματα όπως κατήγγυλαν πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις και η ομάδα μου έχει υποβάλει τροπολογίες που έχουν στόχο τη βελτίωση του κειμένου. Οι τροπολογίες αναφέρονται σημαντικά θέματα πιο συγκεκριμένα διαφύλαξη του συστήματος συλλογής online των στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθήσει νομοθετικά το θέμα σύμφωνα με το άρθρο 11 της Συνθήκης που θα επιτρέπει στις πρωτοβουλίε των πολιτών να μπορούν να προτείνουν τροποποίηση ε, ισχυουσών νομοθετικών προτάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία μέσω ονομαστικής ψηφοφορία η οποία τώρα ξεκινάει. Τέλος. Απορρίπτεται, οπότε τροπολογία 61, ονομαστική ψηφοφορία, ξεκινάει. Τέλος. εγκρίνεται. Άρα το Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει την πρώτη του ανάγνωση. Επόμενη έκθεση για την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών. Η κυρία Μόσκα και ο κύριος Ντόλτον. Κύριε Ντόλτον, νομίζω ότι θέλετε κάτι να πείτε, θέλετε το λόγο, όχι. Α, λάθος έκανα. Ας πάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 97, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Πέρας. εγκρίνεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση. Πάμε στην έκθεση Μπρέσο Βίλαντ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Λεμπρετών έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του εσωτερικού κανονισμού ζητώ οι τροπολογίες να ψηφιστούν και θα ήθελα η τροπολογία μου να ψηφιστεί, να εξεταστεί με ονομαστική ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε την πρόταση του κύριου λοιπόν. Δεν το έχω εδώ. Δεν είχαμε έτοιμα εγκαίρως για, για δομαστική, για να τα συσχυρώσει υπέρ της προτάσης του κυρίου Λεμπρετών. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οπότε πάμε και στις τροπολογίες. Ήταν πολύ ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Πάμε στην τροπολογία 6. Σας παρακαλώ, μη φωνάζετε. Ας ελέγξουμε λοιπόν, γιατί ξέρουμε το αποτέλεσμα. Ας είμαστε δίκαιοι. Καλώς. Έλεγχος. Για την πρόταση Le Ξεκινάει Ξεκινά έλεγχος, τελείωσε ο έλεγχος. Δεν νομίζω ότι θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Ξέρω ότι φοράω γυαλιά, αλλά τα μάτια μου δεν είναι και τόσο άσχημα σε κατάσταση. Λοιπόν, ονομαστική ψηφοφορία για το 6. Πέρας. Εγκρίνεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ολοκληρώνει την πρώτη ανάγνωση. Προχωράμε και απάμε απειλέ κατά τη ασφαλεία που συνδέονται με αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία τη Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενδεχόμενη ανάληψη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωσή του. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Πάμε στην έκθεση Καλνιέται. Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία. Ε, τροπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλο. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφο 7. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλο. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλος. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9 το αρχικού κειμένο, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Παρακαλώ. Για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 1. Ξεκινάει ο έλεγχος. Τέλος. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει συνεπώ. Παράγραφος 30 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλος.